γραπτη Γραπτή δήλωση υπαριθμών 4-2015 για την εγκαθίδρυση ενός Ευρωπαϊκού έτους για την καταπολέμηση της βίας κατά των ε, γυναικών που υπέβαλαν ο συνάδελφος Ταραμπέλα και τα καταθέσα άλλοι βουλευτές. ή 413 διαφορετικές υπογραφές σημαίνει η προψηφία των ε, μελών που απαρτίζουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δημοσιευθεί λοιπόν η σχετική γραπτή δήλωση με τα ονόματα των υπογραφόντων. Την Τετάρτη με βάση το άρθρο 78 του κανονισμού μας σε ε, κοινή πράξη με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου θα υπογράψει